Εσείς σας παρακαλώ πολύ και πάλι για λίγο την προσοχή σας. Όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια της 16ης Ιουλίου ο ε, συνάδελφος Ευρωβουλευτής Κόρβιν Μίκελ ε, προέβησε δηλώσεις ε, οι οποίες δεν συνάδουν με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ρατσιστικής φύσεως παρατηρήσεις και σχόλια. Ε, έλεγξα και ξαναδιάβασα τα πρακτικά αυτή της συνεδρίασης και ζήτησα εξηγήσει από τον κύριο Κόρβιν Νίκελ. Τον παρακάλεσα να διορθώσει τις δηλώσεις του σε να ζητήσει συγγνώμη. Ε, στις 9 Σεπτεμβρίου συναντηθήκαμε κατηδίαν και αρνήθηκε και επιμένει στη θέση του. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δεσμευμένοι να μην προβαίνουν σε δηλώσεις ε, οι οποίες προσβάλλουν σε ανθρώπους είναι ρατσιστικού ή φλετικού περιεχομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού. Κατόπιν τούτου κατέληξα στην απόφαση να επιβάλλω στον κύριο Κόπιν Μίκε μία κύρωση την αφαίρεση 10 ημερήσεων αμοιβών τις οποίες και του τις αφαιρώ, του τις στερώ. Ο συνάδελφος μπορεί βέβαια μέσα σε 14 ημέρες από τώρα, από αυτή τη στιγμή, να ε, καταθέσει έφεση και κατόπιν θα κληθώ εγώ να αποφασίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.